Good morning, everyone. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ε, Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της μεσημερίσης διάταξης, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ όλοι συμφωνούμε και περνάμε γρήγορα στη δημόσια ακρόαση με τους κοινωνικούς εταίρους για τον ρόλο της ε, Τρόικας, ε, Επιτροπή, ΕΚΤ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμπεριλαμβανομένων των πτυχών κοινωνικής, των κοινωνικών πτυχών και των πτυχών της απασχόλησης. Θα συμμετέχει ο κύριος Βότσον, επικεφαλής του Business Europe και η κυρία Νίλσον, γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδικάτων. Θα δώσω το λόγο και στους δύο προσκεκλημένους μας. Πρώτα στην κυρία Βερόνικα Νίλσον για 7 λεπτά και στη συνέχεια στον κύριο Βότσον για άλλα 7 λεπτά. Ναι, βεβαίως ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για κοινή ακρόαση των δύο επιτροπών, γι' αυτό και έχουμε και την χαρά να είμαστε εδώ να συμπροεδρεύουμε την κυρία Μπέρες κοινή συνεδρία τη Επιτροπή τη Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Δίνω το λόγο στην κυρία Νίλσον για 7 λεπτά. Ε, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σα. Ε, μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ. εδώ Εμεί στην ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων θεωρούμε πω η έκθεση που συντάσσεται είναι εξαιρετικά σημαντική και οι δύο γνωμοδοτήσει των δύο επιτροπών περιγράφουν πολύ καλά πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με τι επεμβάσει τη Τρόικα και δείχνουν σαφώ πως οι ενέργειες της Τρόικα δεν είναι συμβατές με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ξέρω πως έχετε εργαστεί πολύ από αυτού και έχετε στείλει και ερωτηματολόγια στα διάφορα ευρωπαϊκά ε, όργανα και οργανισμούς και ούτω καθεξής. Και εμείς το ίδιο κάναμε. Στείλαμε μια, ένα ερωτηματολόγιο στις ενώσεις μας από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία για να συλλέξουμε τις απόψεις τους για να σας δώσουμε τις απαντήσεις μας και εμείς σήμερα. Και επί τη βάση των δικών τους απαντήσεων συντάξαμε μια έκθεση την οποία αποκαλούμε λειτουργία της Τρόικα, την έκθεση του ε, ε, ETUC. Εάν ε, σας ενδιαφέρει, έχω βάλει αντίτυπα εκεί στο τραπέζι και σας παρακαλώ να πάρετε κι εσείς ένα αντίτυπο. Κατά τη γνώμη μας, Αναμφίβολα τα μέτρα λιτότητας που επευλήθησαν από την Τρόικα ήταν εξαιρετικά ευρία και μπορούν να δεχτούν επικρίσεις επί διαφόρων βάσεων. Καταρχήν το ρυθμό της δημοσιονομικής εξηγήνσης, αλλά και ε, το ότι έχουν εστιάσει υπερβολικά στη πτυχή των ε, εισοδημάτων. Μη σεβασμός του κοινωνικού διαλόγου ούτε των κανονισμών για τις εργασιακές αγορές καθώς και ε, των κοινωνικών συστημάτων είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς η Τρόικα αντιμετώπισε τους κοινωνικούς εταίρους. Οι, τα μέλη μας ε, τόνισαν ότι αν και προσκλήθηκαν στις συναντήσεις, αν και στην Κύπρο μόνο σε δύο προσεκλήθησαν, ενώ έγιναν πολύ περισσότερες ε, συσκέψεις με τους εργοδότες, παρόλα αυτά η ποιότητα του διαλόγου ήταν εξαιρετικά φτωχή. Δεν υπήρξε πραγματικός διάλογος, αλλά βασικά επίσημες ε, συσκέψεις που καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι, απλά επειδή είναι υποχρεωμένοι να τους καλέσουν, ενώ οι επαφή δεν έχει πραγματικά νόημα. Οι κοινωνικοί εταίροι, όπω ίσω γνωρίζετε, σε διάφορε χώρε, προσπάθησαν να αναλάβουν την ευθύνη, αν και η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη και όταν ε, πετέφθησαν συμφωνίε δεν έγιναν σεβαστέ από την Τρόικα, Όπω για παράδειγμα η τριμερή συμφωνία που επετέχθη στην Πορτογαλία για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση τον Ιανουάριο του 2012. Αυτή η συμφωνία συμπεριλάμβανε σαφή υποχρέωση για προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ωστόσο η Τρόικα αποφάσισε να περιορίσει τις νομικές ε, ε, ε, επιπτώσεις της συλλογική διαπραγμάτευσης, πράγμα που είχε σοβαρές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στην Πορτογαλία και σε αυτό θα επανέλθω αργότερα. Παρόμοιο συνέβη στην Ελλάδα. Παλαιότερα το ελάχιστο ημερομίσθιο οριζόταν από μια εθνική συλλογική σύμβαση, αλλά το Φεβρουάριο του 2012 η κυβέρνηση υπό μεγάλη πίεση από την Τρόικα περιέκοψε κατά 22% τη ελάχιστα ημερομίσθια και ακόμη περισσότερο για τους νέους εργαζόμενους χρόνους όπου το περιόρισαν κατά 32% ε, και ε, συγκεκριμένα περιόρισαν τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων να ορίζουν τα ελάχιστα ημερομίσθια. Στην Ελλάδα ολόκληρο το σύστημα των ελεύθερων ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει κατακαιρματιστεί. Οι εθνικές και οι τομεακές κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις καταργήθηκαν και σαν να μην έφτανε αυτό η αρχή της συλλογικής εκπροσώπησης δεν ε, υποστηρίζεται πλέον διότι το δικαίωμα για σύναψη κλαδικών συμφωνιών με λιγότερο ευνοϊκούς όρους έχει επεκταθεί στις ε, σε, σε, υπο, σε, σε αποκαλούμενες ενώσεις ή οργανώσεις οι οποίες καταργούνται μόλις ε, επιτύχουν το στόχο τους να, να περικόψουν δηλαδή τα ημερομίσθια. Σύμφωνα με ε, τον Ελληνικό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και διατησίας οι διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές σχεδόν έπαψαν και ε, οι, οι, οι, οι ενισχύ συλλογικές διαπραγματεύσεις μειώνονται σημαντικά. Στην Πορτογαλία ο αριθμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων επίσης ε, ε, περιορίζεται ε, γρήγορα λόγω των πολιτικών που έχουν επιβληθεί εδώ βλέπουμε την μη ανανέωση συλλογικών διαπραγματεύσεων, αυστηρότερα κριτήρια για την παράταση συμφωνιών και την κίνηση προς μια διαδικασία μακριά από τα συνδικάτα, όπου πλέον δεν διαπραγματεύονται τα συνδικάτα εξ ονόματος των εργαζομένων, αλλά διάφορες ενώσεις και συμβούλοι εργαζομένων. Στην Πορτογαλία το 2010, 116 συμφωνίες παρατάθηκαν νομικώς, ενώ το 2013 μόνο 9 ε, τέτοιες συμφωνίες ε, παρατάθηκαν. Πολύ λίγε δηλαδή. Κατά συνέπεια, ο αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από τι συλλογικέ αυτέ συμφωνίε έχει μειωθεί σημαντικά. Στο ιδιωτικό τομέα, πριν την άφηξη τη Τρόικα, 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι καλύπτονταν, ενώ τώρα καλύπτονται μόνο 300.000 εργαζόμενοι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δραματικέ ήταν αυτέ οι αλλαγέ. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των πολιτικών, διότι το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Υπάρχει άνευ προηγουμένου ανεργία σε αυτές τις χώρες, όπως γνωρίζετε, πάνω από το 25% στην Ελλάδα. Στην Πορτογαλία σχεδόν 800.000 θέσεις απασχόλησης, 15% δηλαδή της απασχόλησης έχουν απολεστεί από το 2008. Βλέπουμε επιτεχεινόμενα να αυξάνεται το δημόσιο χρέος στην Πορτογαλία, έχει αυξηθεί από το 94% το ΑΕΠ το 2010 στο 28% και στην Ελλάδα τώρα είναι το χρέος το 176% του ΑΕΠ, αυξημένη φτώχεια λόγω των περικοπών στα ημερομίσθια και στους μισθούς, 17% έχουν πέσει οι μισθοί, οι περιορισμοί στις συντάξεις, στα κοινωνικά επιδόματα, στην κοινωνική πρόνοια και ούτω καθεξής. Μπορώ να, το, μπορώ να πω περισσότερα, αλλά πραγματικά είναι καταθλιπτικό αυτό και απογοητευτικό αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Και δεν είναι εντυπωσιακό ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις κυβερνήσεις τους και στη δημοκρατία εν γέννη, πράγμα που μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τις διάφορες δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου. Να τονίσω και να υπογραμμίσω επίσης ότι αν και η Τρόικα δεν έχει κανένα νομικό καθεστώς, η Κομισιόν και η ΕΚΤ δεσμεύονται από τις συνθήκες. Δεν μπορούν να τις αφήνουν κατά μέρος όταν ενεργούν ε, μέσω της Τρόικα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τους μισθούς. Επίσης είναι υποχρεωμένη να σέβεται και να προωθεί τους κοινωνικούς εταίρους και την αυτονομία αυτών. Ωστόσο η Κομισιόν και η ΕΚΤ έχουν επιβάλει μέτρα τα οποία καταστρέφουν το κοινωνικό διάλογο, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και παρεμβαίνουν διαρκώς στην πολιτική διαμόρφωση των μισθών. Η Κομισιόν πλέον δεν ενεργεί ως θεματοφύλακα στις συνθήκες. Επίσης, ορισμένα από τα μέτρα παραβιάζουν τις συμβάσεις του της Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ε, ότι ορισμένα από τα μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα δεν είναι σύμμορφα προς τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Πέρυσι ε, κατέληξαν ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συμβάσεις περί κοινωνικής ασφάλισης λόγω των μαζικών ε, μειώσεων των των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. Ε, ήγηκε πλέον η ώρα νομικώ να αμφισβητήσει την Κομισιόν και την Έκτη του Ευρωκοινοβούλιο και θα θέλαμε πραγματικά να σας παρακαλέσουμε να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το γεγονός ότι έχετε προνομιακό στάτου ε, μπορείτε εύκολα να φέρετε μια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης έχουμε εκθέσει διάφορες προτάσεις και συστάσεις στην εκθεσή μου. Ξέρω πως έχει ολοκληρωθεί εδώ ο χρόνος μου και δεν θα σας αναλύσω όλες μας τις προτάσεις. Απλά θα κλείσω λέγοντας πως ε, ε, θα θέλαμε αυτή η έκθεση να είναι ένα πρώτο βήμα, ότι θα προβείτε σε μέτρο ώστε να εξασφαλίσετε πως το ό,τι έχει συμβεί μέσω της Τρόικας σε αυτές τις τέσσερις χώρες δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νίλσον. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Watson από το Business Europe, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που καλέσατε την Business Europe να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση και να σας δώσει τις εμπειρίες της από τον, ε, τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να πω ότι Έχουμε επωφεληθεί πολύ από τις παρατηρήσεις των μελών μας, ομοσπονδιών, της Ιρλανδίας, της ε, Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα αναπτύξω σε τρεις τομείς την τοποθέτησή μου. Καταρχάς κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το ρόλο της Τρόικα και μετά θα αναφερθώ στη γενική στρατηγική της ε, Τρόικος προς την ε, υλοποίηση του προγράμματος των προγραμμάτων ανάλογα με τις χώρες με κάποια παραδείγματα και μετά τη διαδικασία της κυβέρνηση. Ως προς το ρόλο της Τρόικα, η Business Europe καλωσορίζει τη θέσπιση της και την υποστήριξη που έχει προσφέρει στις χώρες του, που έχουν ταχθεί στα προγράμματα. Όπως και η Βιρόνικα Νίλσον υπεγράμμισε, είναι σαφές ότι ήταν μεγάλες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτές και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, κυρίως των νέων, που συνεχίζονται, αποτελούν ε, μια πολύ, σημαντική πηγή ανησυχίας. Πλην όμως, θεωρούμε επίσης ότι ήταν αναπόφευκτες οι δύσκολες επιλογές. Σε μερικές περιπτώσεις καθυστέρησαν σημαντικά να ληφθούν και απεδείχθη σε πολλές περιπτώσεις ήταν και απαραίτητε. Και ενώ ήταν συνδεδεμένα τα δάνεια με πολύ σκληρές συνθήκες, πρέπει να υπενθυμίζουμε πάντα ότι η Τρόικα, διακόπτει ο μιλητής, συνεχίστε. Πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η Τρόικα ανέλαβε καθήκοντα σε μια χρονική στιγμή όπου οι περισσότεροι δανειστέ, οι ήταν απρόθυμοι να δανείσουν χρήματα στι χώρε γιατί ήταν πολύ επικίνδυνη η ε, η ανάληψη αυτή τη ευθύνη του δανεισμού και επομένω δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αγορέ οι χώρες. Και έτσι συγκράτησε η παρεμβάση τη της ε, ε, την επέκταση και μετάδοση του προβλήματο γενικότερα στον χώρο του ευρώ και πολύ σημαντικότερους κινδύνους στις χώρες αυτές. Βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπήρξαν προβλήματα προ προς την επεμβάση της Τρόικα. Η κατάσταση όπως είπα στην αρχή ήταν δύσκολη εξ αρχής και έχει οδηγήσει σε σημαντικές και ανησυχητικές κοινωνικές επιπτώσεις η κρίση. Υποτιμήθηκαν οι συνέπειες στην πραγματική οικονομία ορισμένων μέτρων και το ότι τα, οι συνέπειε των μέτρων αυτών δεν επιμερίστηκαν ισότιμα. Ωστόσο, στο βαθμό που υλοποιήθηκαν τα μέτρα, ε, θα δώσουν αποτελέσματα πραγματικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όχι βράχυπρόθεσμα, αν και ήδη βλέπουμε κάποια αποτελέσματα όπως τον περιορισμό των δημοσίων ελλημάτων με πρωτογενές πλεόνασμα για την Ελλάδα όπως προβλέπεται το 2013 συγκεκριμένα. Βλέπουμε τη συμμετοχή τους στις εξαγωγικές, ε, στο εξαγωγικό εμπόριο να αυξάνεται, να μειώνεται το, εργα... το κόστος του εργατικού δυναμικού, όπως παραδείγματι στην Πορτογαλία έχουμε την τελευταία πενταετία την εξέλιξη αυτή, περιορισμό κατά έως 10%, ε, περιορισμό μάλλον ε, σημαντικό της, του ελλείμματος των 10% το 2010 στην Πορτογαλία που τώρα αρχίζει να παίρνει θετικό πρόσημο σιγά σιγά και στην Ελλάδα βλέπουμε αντίστοιχε βελτιώσεις στους στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Η Ιρλανδία έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμά τη, επανέρχεται στην ανάπτυξη, ανακτά την πρόσβαση στις αγορές των κρατικών ομολόγων, όπως άλλωστε και όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από την δημοπρασία Ιρλανδικών ομολόγων. Μπορεί λοιπόν να μην έχουν όλα τα κράτη επανέλθει στις αγορές όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κύπρος, αλλά περιμένουμε ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία το 2014 θα ξαναμπούν στις αγορές, αλλά όπως είπαμε τα επίπεδα της αλλεργίας παραμένουν στις χώρες αυτές πολύ υψηλά, ε, στο και αν παρουσιάσουν κάποια τάση σταθεροποίησης, τα ποσοστά τους παραμένουν πολύ ψηλά. Ως προς τη γενική στρατηγική που υιοθέτησε η Τρόικα και τους στόχους που προσδιορίσε, οι ομοσπονδίες μέλη της Business Europe συμφωνούν εν γέννη με τις στρατηγικές αυτές, υπογραμμίζοντας πάντα ότι η ε, σταθεροποίηση της, της οικονομικής κατάστασης, εξυγέννηση του προϋπολογισμού, περιορισμός των δαπανών χωρίς αυξήσεις της, ε, ε, τις δαπάνες είναι όροι για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της οικονομίας. Αν και θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στις υποδομές, παραδείγματι αυτές των, των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ε, κάποια προβλήματα εντοπίζονται ως προς την υλοποίηση των προγραμμάτων, εκεί όπου αυτή δεν ήταν πάντοτε επαρκώς εξισορροπημένη, γιατί ε, δινόταν προσθέτει έμφαση σε κάποια στοιχεία των προγραμμάτων, ενώ παραγνωρίζονταν κάποια άλλα. Στην Ελλάδα, επί παραδείγματι, ήταν δυσανάλογη η προσοχή που δόθηκε ως προς την ε, ίσπραξη φόρων, ή την επιβολή φόρων καλύτερα, ενώ δεν δόθηκε επαρκή έμφαση ω προ τι μεταρρυθμίσει που θα περιόριζαν τι δαπάνε του δημόσιου τομέα ή θα οδηγούσαν στη μεταρρύθμιση σε διάφορου επαγγελματικού κλάδου ε, και στην παραγωγική οικονομία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε εσωτερικέ πολιτικέ αντιστάσει στην ελληνική ε, περίπτωση ε, ίσως θα μπορούσαν να σκεφτούν περισσότερες πιέσεις όπως, όπως πιστεύουν οι ομοσπονδίες μας για πιο διαρθρωτικές αλλαγές. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας η Τρόικα αλλά και οι ομοσπονδίες μέλη μας θεωρούν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα από την εξυγίανση των δημοσιονομικών ε, ίσως ε, να μην υλοποιήθηκαν ακριβώς οι προβλέψεις, αλλά πάνω απ' όλα ανησυχεί η Ομοσπονδία μέλος ως προς την ταχύτητα αντίδρασης της Τρόικας όταν είδε ότι δεν υλοποιούνταν οι προκλήσεις, ότι δηλαδή δεν ήταν επαρκώς ταχεία η αντίδραση της Τρόικα για να προσαρμόσει το πρόγραμμά της στις συνθήκες. Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της απομόχλευσης των τραπεζών στην Πορτογαλία, με το επίπεδο των πιστώσεων που αναπτύχθηκαν στο μακροοικονομικό πλαίσιο, πράγμα το οποίο επηρέασε τις δυνατότητες δανεισμού πολλών επιχειρήσεων. Για την Κύπρο, η Ομοσπονδία μέλο θεωρεί ότι εν γέννη είναι ευπρόσδεκτη η παρέμβαση τη Τρόικα με μια προσπάθεια για αλλαγή και κυρίω οι μεταρρυθμίσει που έχουν να κάνουν με την πραγματική οικονομία βαίνουν προ την ορθή κατεύθυνση με περιορισμό στον όγκο του δημόσιου τομέα, των δαπανών των κρατικών, της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε... Ε, μπορεί ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία της Κύπρου να καθυστερήσει ακόμη. Υπάρχουν όμως μέσα μεταφοράς ή μετακύλησης του βάρους ιδιαίτερα ως προς τις ε, τράπεζες οι οποίες παρουσίασαν προβλήματα. Ε, μετακύληση του βάρους λοιπόν προς τους επενδυτές οι οποίοι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο. Άρα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η Ομοσπονδία πάντως από την Κύπρο μας λέει ότι ήταν πολύ σημαντική η επιβάρυνση που στην οποία οδήγησε αυτή η μετακύληση και ως εκ τούτου χάθηκε σημαντικό κομμάτι ρευστότητας από την αγορά, την επιχειρηματική. Για την Ιρλανδία επίσης υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, πιο περιορισμένες αυτή τη φορά οι οποίες πάντως ακολουθούν υφιστάμενα ε, σχέδια της κυβέρνησης για την δημοσιονομική εξυγένση. Για να ολοκληρώνω λοιπόν, μια και δεν έχω χρόνο, στο θέμα της διακυβέρνησης, η Τρόικα ήταν ασφαλώς μια προσωρινή ρύθμιση, μια λύση προσωρινή που εξευρέθησε σε περίοδο κρίσης και ως εκ τούτου είναι σχεδόν φυσιολογικό το ότι υπήρξαν προβλήματα Γι' αυτό άλλωστε είναι και σημαντική πολύ αυτή η συνεδρίαση ώστε να εντοπιστούν οι λύσεις και οι δυνατότητες για βελτίωση αν τυχόν εμφανιστεί τέτοιο πρόβλημα πάλι στην Ευρώπη, τουλάχιστον να διδαχθούμε από τα λάθη που έγιναν. Και ίσως θα πρέπει να προσθέσω ότι σε ένα-δύο χρόνια όταν έχουν κλείσει όλα τα προγράμματα όπως ελπίζουμε τη Τρόικα θα ήταν σκόπιμο να ξανακοιτάξουμε με πιο ψύχρεμο μάτι και να αξιολογήσουμε πάλι το τι έχουμε διδαχθεί από την εμπειρία αυτή. Για τη διαφάνεια δεν ήταν ε, πολύ ε, ορατή οι, ορατές οι επιλογές αυτές, διαφάνεια δηλαδή δεν υπήρξε. Αν θέλετε να κλείνω μάλιστα. Ένα πράγμα θέλω να επισημάνω σε αυτό που είπε η Βερόνικα για την εμπλοκή των επιχειρήσεων, γιατί υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις ε, είχαν επαφή και εμπλοκή στη λήψη των αποφάσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και έχοντας εκπροσωπήσει και εγώ στο παρελθόν συνδικάτα αντιλαμβάνομαι ότι η Βερόνικα θεωρεί πως μπορεί να έγιναν πολλές συνεδριάσεις αλλά δεν έδωσαν αποτελέσματα. Σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βότσον. Τώρα αρχίζει η συζήτηση. Τρία λεπτά. Ο εισηγητής από το ΕΛΚ. Τρία λεπτά ο εισηγητής από τους σοσιαλιστές και 4,5 λεπτά ο εισηγητής Αλεχάνδρο Θέρκας από την Επιτροπή Οικονομικών. Ο κύριος Καράς είναι ο εισηγητής του ΕΛΚ Δεν μπορεί να είναι εδώ όμως, οπότε θα πάρω εγώ τον λόγο ανταυτόν. Πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Κάρας, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει εδώ σήμερα. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι ο κύριος Καράς στο σχέδιο εκθεσής του επιμένει για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Ο κύριος Κάρας λοιπόν θέλει να ρωτήσει σε τι βαθμό οι εθνικές κυβερνήσεις είχαν διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους προτού οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Άλλη ερώτηση. Έχει να κάνει και με την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου στις διάφορες χώρες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις βασικά που έχει ο κύριος Κάρας, ο εισηγητής του ΕΛΚ. Θα δώσω τώρα το λόγο για τρία λεπτά στον κύριο Λία ο οποίος είναι ο εισηγητής των σοσιαλιστών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Παύλο. Λυπάμαι που ο συνάδελφος Κάρας δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν ξέρω γιατί η Δεν νομίζω ότι επειδή αγνοεί η ομάδα του την κοινωνική διάσταση που δεν βρίσκεται εδώ, γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Λοιπόν, θα αρχίσω με τα συνδικάτα. Ρωτάω λοιπόν, Θα μπορούσε η εργοδοσία, η οποία δεν συμφωνεί βέβαια με τις δικές σας θέσεις, να σας πει ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας στις χώρες μνημονίων δεν αντέχουν πια και πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Τι έχετε να πείτε σε αυτό. Δεύτερον, κάποιοι λένε ότι σε αυτές τις χώρες υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Πιστεύετε κι εσείς ότι υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας Και άρα πρέπει να πέσει το κόστος εργασίας, όπως λέει η Τρόικα. Τρίτον, γνωρίζετε να υπάρχουν μελέτες που να κάνουν αυτή τη σχέση, δηλαδή αύξηση των ανισοτήτων, η μείωση των ανισοτήτων ευνοεί ή όχι την ανάπτυξη. Αυτά για τα συνδικάτα. Τώρα, για την εργοδοσία και τον εκπρόσωπό της. Στην σημερινή μας ακρόαση δεν συμφωνείτε βέβαια με την εκπρόσωπο των συνδικάτων. Είναι σημαντικό πράγματι να έχουμε και τις δύο απόψεις, και τον με και τον δε. Οπότε θέλω και εσάς να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Τα Πράγματα που θα μπορούσαν να σας ρωτήσουν τα συνδικάτα, αλλά σας τα ρωτάω κι εγώ. Μελέτες του ΟΣΑ πρώτα απ' όλα προοπτικές απασχόλησης. Δεν υπάρχει εκεί σχέση ανάμεσα στην προστατευτική νομοθεσία για την απασχόληση και τις οικονομικές επιδόσεις των διαφόρων χωρών. Ενώ εσείς μιλάτε για διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και κυρίως στο δίκαιο εργασίας, στο εργασιακό δίκαιο. Μπορείτε να δικαιολογήσετε την ε, τοποθέτησή σας αυτή. Δεύτερη ερώτηση για το κόστος ε, εργασίας. Έχω δουλέψει πολύ πάνω στο πρόβλημα αυτό όταν ήμουνα στο πανεπιστήμιο μάλιστα. Και από όσο γνωρίζω είναι πολύ επίμαχο το θέμα ε, μισθή αν πρέπει να μειώνονται ή όχι και οι οικονομολόγοι προβληματίζονται πολύ και διαφωνούν μεταξύ τους σχετικά με το κόστος εργασίας και τους μισθούς. Εσείς σε ποιες μελέτες βασίζεστε για να δικαιολογήσετε τις μεταρρυθμίσεις που προτείνετε για το κόστος εργασίας. Και τέλος, για τους ε, δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Εσείς που είσαστε ειδικοί της εργοδοσίας, έχετε κάποια άποψη για τις πρόσφατες μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τους ε, πολλαπλασιαστές. Ο κύριος Μπλανσάρ ξαναείδε τις μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είπε ότι είναι μάλλον πάνω από 1,5. Εσείς σε τι τιμή καταλήγετε και έχει αυτό επιπτώσεις στις μεταρρυθμίσεις που προτείνεται για την μείωση των δημοσίων δαπανών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Λιάμ. Τώρα, εκ μέρου της Επιτροπής Απασχόλησης, το λόγο έχει ο εισηγητής της για 4,5 λεπτά. Παρακαλώ κύριε Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, αγαπητοί προσκεκλημένοι εδώ στην ακρόασή μας, Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας. Είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας εδώ ακριβώς για να καταλάβουμε καλύτερα ένα μέρος του προβλήματος το οποίο κινδυνεύει να μείνει στη σκιά. Χρησιμοποιούμε το χρόνο μας όσο καλύτερα μπορούμε για τα μακροοικονομικά, τα δημοσιονομικά. Μερικές φορές ξεχνάμε όμως ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα κλαμπ τραπεζιτών, ούτε μια οικονομική καθαρά οντότητα. Όχι, όπως λένε και οι συνθήκες, είναι κυρίως στην υπηρεσία των πολιτών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την Επιτροπή Απασχόλησης στις συζητήσεις αυτές. Τι επιπτώσεις λοιπόν είχαν τα προγράμματα αυτά στις τέσσερις χώρες που εφαρμόστηκαν στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Τι έγινε με την απασχόλησή τους, στα σχολιά τους, στα παιδιά τους, στο μέλλον τους. Τι συνέβη αυτά τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν στην Επιτροπή Απασχόλησης ετοιμάζουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Εγώ έχω ήδη ετοιμάσει το σχέδιο. 250 τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Συζητάμε με το κοινό. Παίρνουμε πάρα πολλά έγγραφα από πανεπιστήμια, από κέντρα μελετών. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έγιναν μελέτες σε βάθος για τις κοινωνικές συνέπειες της παρουσίας της Τρόικα. Όλα αυτά εμπλουτίζουν βέβαια τις γνώσεις μας για το τι ακριβώς συνέβη. Θέλουμε να κάνουμε μια πλήρη ανάλυση για τις συνέπειες και για το μέλλον, γιατί δεν είναι δυνατόν να μένουν θέματα σε κρεμότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα μελετήσουμε τρία κυρίως στοιχεία. Πρώτον, επιπτώσεις στους τρεις κοινωνικούς στόχους στρατηγικής 2020 και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση προς εσάς. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά, πιο μακριά δυσκολεύονται οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουμε μια Ευρώπη αριστείας και να αντιμετωπιστεί η κρίση. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε την τάση να κοιτάμε βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Δεύτερη ερώτηση για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Και η διεθνής διάσταση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Μέχρι τώρα έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πλήττουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων επειδή έχουμε λιτότητα ή άλλα πράγματα τα οποία στο κάτω-κάτω έχουν ψηφιστεί και με δημοψήφισμα στις χώρες μέλη. Τι γίνεται λοιπόν με τις συστάσεις αυτές, έχουν τηρηθεί ή δεν έχουν τηρηθεί οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνθήκες που έχουν οδηγήσει στα, στη χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα ή άλλα πράγματα που έχουμε υπογράψει από το Εθνές Γραφείο Εργασίας κλπ. Εμείς θα λέμε και τα λέμε. Υπάρχει η Σύμβαση 27, τα συνδικαλιστικά, η Συλλογική Σύμβαση, η Ελάχιστη Μισθή κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα θέλω να ξέρω έχουν γίνει σεβαστά, έχουν τηρηθεί ή όχι. Πρέπει να το ξέρει η κοινή γνώμη. Έπειτα για τις συστάσεις για το μέλλον. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις επικρίσεις που ακούγονται και να λάβουμε υπόψη μας τι έγινε. Μέχρι τώρα όλα είχαν γίνει καλά. Αν αυτή είναι η απάντηση, ε, θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Τι νόημα τότε έχει η πολιτική. Εμείς, αντίθετα, θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον και να δούμε τι θα αλλάξουμε στο μέλλον. Οπότε, θέλω να ρωτήσω τώρα πιο συγκεκριμένα. Τα συνδικάτα δεν μίλησαν για τις δημόσιες υπηρεσίες. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία. Τι γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση. Τι λένε τα μέλη των συνδικάτων σας για τις επιπτώσεις που είχαν αυτά τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητά τους. Έπειτα, στα πλαίσια του κοινωνικού τριμερούς διαλόγου, μερικές φορές υπήρξε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων, υπήρξαν συζητήσεις με τους επιτρόπους, με τον Όλυ με την Τρόικα, με το Eurogroup, με το Εκοφίν οι κοινωνικοί εταίροι, τα συνδικάτα ή και οι Europe Business ρώτησαν ε, τους ε, ανθρώπους αυτούς, τους μίλησαν μαζί τους. Έπειτα, κάποια πράγματα για τα οποία δεν άκουσα να μιλέτε. Σε τι βαθμό καταστράφηκαν επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πήγαμε στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία βέβαια. Οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε μεγάλη αγωνία γιατί νιώθουν ότι καταστρέφεται ο επιχειρηματικός ιστός στις χώρες. Έχουν χαθεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Έχω 30 δευτερόλεπτα πρόεδρε, με κόβετε ακόμα. Α, τι πέρασαν, ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο ερωτήσεις μου και ελπίζω μετά να μου δοθεί ευκαιρία να ξαναπάρω το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Θέρκας. Τώρα. Η κυρία Νίλσον για να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας, κύριε Νίλσον. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ε, αρκετά δύσκολες ορισμένες εξ αυτών. Θα, θα ξεκινήσω με το ερώτημα του πρώτου ε, παρεμβαίνοντα. Ε, κοιτάξτε, του κυρίου Κάρας θα το, το λιγότερο που θα περίμενε κανεί είναι να γίνονται σεβαστές οι συμφωνίε οι οποίε έχουν συναυθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό ποτέ δεν συνέβη στην Πορτογαλία. Εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα παρότι η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, τότε θα ήλπιζε κανεί και θα ανέμενε ότι θα γίνονταν σεβαστές αυτέ οι συμφωνίε από την Τρόικα και από την κυβέρνηση. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που μπορώ να σα δώσω, αλλά ίσω και να προσθέσω ότι ε, Πολλές ε, κατηγορίες έχουν γίνει, αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε Τρόικα και κυβέρνηση. Η Τρόικα λέει, όχι δεν ήμασταν εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτό που ήθελε, εμείς απλώς ε, προτάσεις κάναμε. Οι κυβερνήσεις λένε, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί μας πίεζε η Τρόικα και πάει λέγοντας. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Έπειτα, για την ανταγωνιστικότητα. Να σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι δεν ήταν κρίση ανταγωνιστικότητας αυτή η κρίση, το ξεκίνησε, που πράγμα που θα μπορούσε κάνει να σκεφτεί ε, όταν ακούει κάποιες παρεμβάσεις. Ε, πρόκειται για τραπεζική κρίση. Ξέρουμε όλοι πω δεν είναι τέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι κάποιο τέλειο δημιούργημα. Οπότε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τρόικα και οι κυβερνήσει είναι να δημιουργήσουν εσωτερική υποτίμηση και αυτό είναι σαφέ. Το πρόβλημα δεν είναι η ανταγωνιστικότητα. Δεν λέω πως αυτές οι χώρες ήταν τέλειες πριν την κρίση. Όχι. τελειότητας δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Τέλεια οικονομία και τέλεια χώρα. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πρόκειται αρχικά για τραπεζική κρίση, η οποία οδήγησε στην κρίση του χρέους. Και αν δούμε και τα αριθμητικά στοιχεία, καθίσατε σαφές πως οι πολιτικές της Τρόικα έχουν αποτύχει. Δεν αύξησαν την ανταγωνιστικότητα σε αυτές τις χώρες. Αυτό που συνέβη είναι πως έχει αυξηθεί η ανεργία, η φτώχεια σε τεράστιο βαθμό. Τα, οι μισθοί έχουν περικοπεί ε, κατά 17% στην Ελλάδα. Ε, έχει μειωθεί το κόστος της εργασίας. Με διαφορετικό τρόπο όμως θα μπορούσε να γίνει, όχι μόνο μέσω της μείωσης των μισθών, εφόσον θεωρείται απαραίτητη αυτού του είδους η πολιτική. Πάντως, δεν είναι αλήθεια πως οι χώρες αυτές κατανάλωναν πέραν από το επίπεδο πρόνοιας και έπειτα γιατί ε, έχουν επιβαρυνθεί οι εργαζόμενοι περισσότερο που σίγουρα δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι για την κρίση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και έπειτα... Μισό λεπτό γιατί δεν είμαι βέβαια ότι ε, έχω σωστά καταγράψει ερωτήσεις σας. Ε, υπάρχει κάποιος διάλογος με την ε, Κομισιόν, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά σε ποιο βαθμό ε, γίνεται αυτό σωστά. Δηλαδή όταν η Κομισιόν αντιπροσωπεύεται στην Τρόικα, πώς φτάνει σε κοινέ θέσεις. είναι όντως αυτή η κοινωνική εταίρεια αντιπροσωπευτική, όντως ε, ε, αντιπροσωπεύουν τους εργαζόμενους στις χώρες τους. Εσείς μπορείτε να τα ξέρετε περισσότερα, καλύτερα, γιατί εσείς έχετε συντάξει αυτές τις νομοδοτήσεις. Πάντως υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σίγουρα εδώ ε, και εμείς θα αναμέναμε η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο να λάβουν μέτρα για αυτό το θέμα. Αυτά έχω να πω. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις θα συνεχίσω και αργότερα. Σας ευχαριστούμε κυρία Νίλσον, ήσασταν και στην ώρα σας, ο κύριος Βότσον. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Στην πρώτη ερώτηση του κυρίου Κάρας για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, νομίζω πως το ανέφερα αυτό στο τέλος της παρέμβασής μου. Υπήρξε συμμετοχή, αλλά θα, ήταν, θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματική η επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους, αν είχαν θεσπιστεί σαφέστερες ε, μερίσεις διατάξεις ε, και αν είχαν ε, τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι από πλευράς της Τρόικας, κάποια μεγαλύτερη τυποποίηση για το δεύτερο σύνολο ερωτήσεις, ερωτήσεων σε σχέση με την αγορά εργασίας. Δεν ε, θα μιλήσω εγώ τώρα αν ήταν ε, κρίση τραπεζική ή κρίση ανταγωνισμού. Απάντως, αυτό που ε, είναι βέβαιο είναι ότι η ανταγωνιστικότητα της εργασίας αυξήθηκε λόγω της κρίσης. Βέβαια, όταν μπαίνει κανείς σε μια νομισματική ένωση, ξέρει πως δεν θα έχει τη δυνατότητα να υποτιμήσει την συναλλαγματική του ισοτιμία. Αυτό παίζει φυσικά στη, στους μισθούς ε, που αυξάνονται σύμφωνα και με την παραγωγικότητα, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Και εκεί που είδαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους μισθούς ε, ενώ προχωρούσαμε προς την κρίση, είδαμε και τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας στις ίδιες χώρες. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν προσαρμογές αγοράς εργασίας. Ε, χρειάζεται οι μοναδιές το μοναδιαίο κόστος μάλλον της εργασίας να πέσει ε, σε κάποιες από τις χώρες ε, των μνημονίων και αρχίζουμε να βλέπουμε τις βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα που ανέφερα στην ε, παρέμβασή μου. Δεν θα μπω, φοβούμαι, στο συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Θα το αφήσω αυτό για τους εμπειρογνώμονες. Απλά να σημειώσουμε ότι βεβαίως υπάρχει ένα αρνητικό ε, βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα όταν μιλάμε για δημοσιονομικούς ε, πολλαπλασιαστές και ότι περνάει χρόνος μέχρι ότου να ξαναβρει την ίδια φόρμα η οικονομία. Τέλος, ε, για να πω και για να τονίσω και σίγουρα δεν είπα ότι η Τρόικα τα έκανε όλα καλά και Άγια. Σίγουρα δεν είπα πως όλα πάνε καλά τώρα, αλλά και μάλιστα ανέφερα το ότι παρότι τα προγράμματα ε, ήταν βασικά οι σωστέ στρατηγικέ, υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την ισορροπία στην εφαρμογή του. Ε, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αναφέρετε το 2020, αν είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση σε σχέση με το Ευρώπη 2020 από ό,τι πριν. Εγώ θα πω το εξή. Εγώ πιστεύω πω η κρίση ε, ήταν μεγάλο εμπόδιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν δει κανεί τα επίπεδα τη ανεργία. Όμω ταυτόχρονα πιστεύω Αντί να σκεφτόμαστε το 2020, περισσότερο αν δούμε την ε, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, είναι βέβαιο ότι ορισμένε από τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που τέθησαν σε εφαρμογή στι ε, χώρε των προγράμματο αλλά και σε άλλε χώρε, ε, και αν σκεφτούμε την Ισπανία και κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας εκεί, αυτέ οι μεταρρυθμίσεις θα εξυπηρετήσουν την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη μακροπρόθεσμα και θα βοηθήσουν στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γουότσον και τώρα θα δώσω το λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Ρωσματικής. και έτσι ερχόμαστε στην ε, παρέμβαση των σκιωδών συγητών, Επιτροπή Απασχόλησης, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κυρία Μπάστος, αντικαθιστά ο κύριος Φερνάντε. Έχετε το λόγο. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, όπω υπόθηκε, η συνάδελφο Ρεζίνα Μπάστο, που είναι σκιώδη εισηγητή τη Επιτροπή Απασχόληση, δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματό τη, πράγμα το οποίο και θα κάνω. Η οικονομική κατάσταση τη Ελλάδα, τη Πορτογαλία, τη Ιρλανδία και τη Κύπρου επιδεινώθηκαν μέσω τη δημοσιονομική χρήση και χρειάστηκε να δοθούν επίγουσε απαντήσει. Χωρί τα προγράμματα προσαρμογή, οι συνέπειε θα ήταν ακόμη πιο σοβαρέ και με περισσότερο κόστος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ωστόσο θα πρέπει να πούμε και να παραδεχτούμε ότι η εφαρμογή των μέτρων των ε, προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής επηρέασαν άμεσα και έμεσα τα επίπεδα απασχόλησης και τις συνθήκες διαβίωσης των ε, πολιτών μας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο στον Ταβός, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Τράκη είπε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία ε, δίνει ε, σήματα ανάκαμψης, οι οικονομικές αγορές άρχισαν να σταθεροποιούνται και ορισμένα κράτη-μέλη ήδη πρόκειται να βγουν σύντομα από, ε, μάλλον ήδη βγήκαν από τα προγράμματα προσαρμογής, Ισπανία και η Ιρλανδία. Μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς διαρθωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Οι χώρες αυτές που έκαναν τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις με στόχο την παραγωγή και την αγορά εργασίας βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την οικονομική ανάκαμψη. Έτσι ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, ε, δεν ξέρουμε αν οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν τα πήγονται αυτά μέτρα ε, θα ενδυναμώσουν την αγορά εργασία και θα ευνοήσουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και τέλο, ποιε είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να σεβαστούμε την εξυγίαση ε, των κρατών μελών, τη δημοσιονομική εξυγίαση και που στη συνέχεια θα επιτρέψουν την οικονομική ανάκαμψη, την κοινωνική δικαιοσύνη και θα υπερασπιστούν και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αν δεν θέλετε να σας διακόπτω, θα παρακαλώ να πηγαίνετε κατευθείαν σε ερωτήσει σας. Οι συνάδελφοι τώρα εκ μέρου των φιλελευθερών δεν είναι παρόντε και έτσι περνώ στην ομάδα των Πρασίνων και δίνω το λόγο εκ μέρου τη Οικονομικής και Ζωματική Επιτροπής στον Φίλιπ ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στα αγγλικά καλύτερα και, και απευθύνομαι στον εκπρόσωπο της Business Europe. Θα μου επιβεβαιώσετε ότι καλύπτουν κατά 25% τον προπολογισμό σας οι τράπεζες. Φαντάζομαι ναι, πολύ καλά. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε για τις τράπεζες, γιατί προφανώς σας άρεσε η δουλειά της Τρόικα, εκτός από το ότι πολλοί επιέμειναν στην φορολογία και λιγότερο στον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Άρα τους στόχους σας τους έχετε επιτύχει και φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένοι, άλλωστε δεν το κρύβετε. Η εξή ερώτηση λοιπόν από μένα. Φαίνεται να μας λέτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς την κατανομή του βάρους. Θα συμφωνήσετε λοιπόν ότι στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Ισπανίας αλλά ασφαλώς και της Ελλάδος, εάν κάποιοι μπόρεσαν να δανειστούν κατά τρόπο ανεύθυνο, αυτό δείχνει ότι υπήρξαν και εκείνοι ε, από την άλλη πλευρά που ήταν διατεθειμένοι να τους δανείσουν κατά τρόπο ανεύθυνο, από τα μέλη σας δηλαδή. Δηλαδή συμφωνείτε ότι θα έπρεπε κάποια από τα μέλη σας να επιβαρυνθούν με ένα μεγαλύτερο μερίδιο του ε, του προβλήματος που οδήγησε τελευταία ανάλυση λόγω του ανεύθυνου δανεισμού στη Φούσκα, στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα ώστε να μην επιβαρυνθούν μόνο αυτοί που βρίσκονται πιο αδύναμοι. Και παρακαλώ να ετοιμάσετε καλά την απάντησή σα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω δει αξιόπιστες απαντήσει από την Business Europe. Από εδώ και μπρο λοιπόν πώ πάμε, πώ προχωρούμε. Για την κυρία Νίλσον θέλω να ρωτήσω το εξή. Ποια διέξοδο βλέπετε από την EDUC, πώς μπορεί να ξαναδοθεί όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, πώς μπορούμε, μια και φαίνεται περισσότερη έμφαση να δίνεται στις κοινωνικές πτυχές στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να λέει η Επιτροπή, πώς μπορούμε τα six-pack και τα δύο-pack, τα two-pack να τα εξορροπήσουμε έτσι ώστε να είναι πιο ισότιμη η διακυβέρνηση, το governance και τι σκοπεύετε να πείτε σε ώψη ενός κοινο, μιας κοινωνικής διάσκεψης κορυφής, γιατί από απαντήσεις συγκεκριμένε δεν έχουμε δει ακόμα. Ευχαριστώ εκ μέρους των Πρασίνων, αλλά αυτή τη φορά εξ ονόματος ε, ε, της Επιτροπής της Επασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της κυρίας Κορνέλης συγκεκριμένα, ο κύριος Γκίγκολτ. Στα αγγλικά. Καταρχάς, θα ήθελα η TUC να μας ε, πει τι είδους συστάσεις έχει, γιατί βλέπω ότι δεν προλάβατε να τις αναπτύξετε. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν μια ανάπτυξη στο θέμα των συστάσεων και επίσης για την Business Europe, διότι εξεπλάγει. Όταν άκουσα από την ETUC ότι υπήρξαν παραβιάσεις στο δίκαιο και η Business Europe από την άλλη δεν επέμεινε καθόλου ως προς το ζήτημα της νομιμότητας. Μπορείτε να σχολιάσετε στις παραβιάσεις αυτές που επικαλείται η TUC. Γιατί φαντάζομαι ότι υπήρξε ανάγκη για εσωτερική υποβάθμιση σε ορισμένες χώρες και αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Από την άλλη, ωστόσο, δεν μπορεί απλά και μόνο να αποφασίσετε ότι θα παραβιαστεί το δίκαιο και ότι αυτή η παραβίαση του δικαίου ε, ε, δικαιολογείται από το σκοπό που επιδιώκεται δεν μπορεί ένα σκοπό να γιάσει μέσα σε ένα κράτο δικαίου. Ναι, και δεν σχολιάστε καθόλου, λοιπόν, θα θέλω τι απόψει σα. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Και τώρα, εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Ζούμπερ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση προς την Business Europe. Θα ήθελα να σχολιάσει τα νούμερα που έχουν να κάνουν με τις αυξανόμενες ανισότητες σε επίπεδο πλούτου. Δηλαδή, η TUC εδώ στο εγγραφό της έχει δώσει στοιχεία για την μείωση του αξίας του μισθού, για παράδειγμα στη χώρα μου συνέβη αυτό, και ενώ ταυτόχρονα η αξία του πλούτου των βασικών ε, εκατομμυριούχων αυξήθηκε. Γιατί σε μια στιγμή όπου όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες, όπως λέει η Τρόικα. Δεύτερο ερώτημα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη χώρα μου, Πορτογαλία, από τη μια πλευρά ω την άλλη τη Πορτογαλίας βλέπουμε μικρομεσαίε επιχειρήσεις ε, και του επιχειρηματίες που είναι απελπισμένοι γιατί κλείνουν συνέχεια τα επιχειρήσει τους. Αυτοί οι μικρομεσαίοι αντιπροσωπεύονται στα λόγια σα, όταν είπατε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος συμφωνεί με τα μέτρα της Τρόικα. Και η άλλη μου ερώτηση πάει προς την ETUC. Ε, Μιλήσατε για την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής ε, ομόνοιας στην Πορτογαλία δεν υπήρχε γιατί η τριμερή συμφωνία απέκλει απλώς το βασικότερο αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο των Πορτογάλων, που δεν, των Πορτογάλων εργαζόμενων που δεν είχε υπογράψει καμιά συμφωνία. Θέλω αυτό μου το σχολιάσετε. Και έπειτα μια τελευταία ερώτηση και προς τους δύο μιλητές. Είναι αλήθεια ότι οι επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους και δεν ήταν έτοιμοι να επενδύσουν. Σε μια δημοκρατία όμως η οικονομική εξουσία είναι αυτή που θα καθορίζει τις πολιτικές ή η πολιτική εξουσία που πρέπει να διαπραγματευτεί με την οικονομία πολιτικές που θα είναι ευνοϊκές για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ξαναδίνω το λόγο στους δύο προσκεκλημένους, αντιστρέφοντας αυτή τη φορά τη σειρά. ξεκινώ με τον κύριο Γότσον, τέσσερα λεπτά και μετά τη Βερόνικα Νίλσον. Και μια και όσοι δικαιούνται να μιλήσουν αυτοδικαίως έχουν ε, μιλήσει. Θα αρχίσουμε μια διαδικασία catch the eye με όποιον ενδιαφέρεται. Έχω σημειώσει ήδη τον κύριο Πουπάκη. Κύριε Βότσον, έχετε το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Βεβαίως. Τα σχόλια του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα τα είχα στηρίξει. Ρωτάτε πώς μπορεί να αρχίσει και πάλι ανάπτυξη στο σημερινό πλαίσιο. Δύο τομείς θα αναφέρω. να συμπληρωθεί η ενιαία αγορά υπηρεσιών και μείωση του διοικητικού άχθους με καλύτερες ρυθμίσεις. Να, δύο τομεί στου οποίου θα έπρεπε να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει παρετέρω ανάπτυξη. Θέλω όμω να επικεντρωθώ λιγάκι στι ερωτήσει του κύριου Λάμπερτ, για παράδειγμα. Δεν ήξερα το στοιχείο αυτό. 25% του προπολογισμού μας έρχεται από τι τράπεζε, λέτε. Δεν το ήξερα. Με πολύ ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσω. Αυτό όμως που δεν συμμετέχουν στην Business Europe οι τράπεζε, ρωτά ο κύριο Λάμπερτ απάντηση του κ. Βότσον. Ναι, υπάρχουν μέλη σε ομοσπονδίες, κάποιοι είναι, έχουν τράπεζες, αλλά αυτό το 25% πολύ ενδιαφέρον είναι, θέλω να το δω. Η ίδια Business Europe μας έχει δώσει το στοιχείο αυτό, λέει ο κύριος Λάμπερτς. Καλά, με ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσω και θα δω, λέει ο κύριος Βότσον. Τώρα λοιπόν για τις τράπεζες. Η Europe Business είναι σαφής ότι χρειάζεται ρύθμιση και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες στο ρυθμιστικό σύστημα το οποίο οδήγησε στην κρίση. Μερικές φορές κάποιες τράπεζες, ναι, δάνεισαν ανεύθυνα. Και καμία αμφιβολία ότι κάποιες από τις τράπεζες αυτές είναι και μέλη μας. Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι θέλουμε βελτιώσεις στο ρυθμιστικό σύστημα ώστε να υπάρξει και πάλι ισορροπία. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, βασικά και νομίζω ότι το είπα και στην αρχή. Ότι δηλαδή οι επενδυτές αναλαμβάνουν τις ευθύνες των επενδυτικών τους αποφάσεων. Οπότε συμφωνώ με ένα πακέτο bail-in, διάσωσης με ίδια μέσα δηλαδή, που υπογραμμίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάσωση που συμμετέχουν οι επενδυτές και αναλαμβάνουν το βάρος αντί για τους φορολογούμενους. Στηρίζω επίσης την Τραπεζική Ένωση. Το κείμενο το στηρίζουμε για να υπάρξει μια εξυγένση, ένα ταμείο εξυγένσης το οποίο θα συμμετέχουν οι τράπεζες. Εδώ συμφωνώ. Τα υπόλοιπα, άμα θέλετε, θα μπορούσαμε με περισσότερες λεπτομέρειες να τα συζητήσουμε διμερώς. Στον κύριο Κίκολτ τώρα. Όντως δεν είπα στην αρχή τα πάντα. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν ήξερα κάποια από τα πράγματα που είπατε για το, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Σίγουρα θα <clears throat> έχει δημοσιευθεί. Εγώ δεν το ήξερα σίγουρα, θα υπάρξουν κάποιες παραβιάσεις, αλλά οι, τα μέλη μας δεν θέλουν να παραβιάζεται η νομοθεσία. Είμαστε υπεύθυνε επιχειρήσεις. Και τέλος, όσον αφορά τις ανισότητες και την κατανομή του πλούτου, εδώ θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε τόσο υψηλά επίπεδα ανισότητας είναι επειδή έχουμε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα ε, ανεργίας και γι' αυτό και εμείς θέλουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την απασχόληση και ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων. Πιστεύουμε ότι χρειάζονται μέτρα όπως αυτά που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις ανισότητες. Κύριος Λάμπερ, ο κύριος Γιγόλτ μάλλον. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Στην ΕΚΟΝ έχουμε την ε, συνήθεια, αν κάποιος δεν απαντήσει, να μπορούμε να επανέλθουμε. Ναι, όταν είναι η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα, λέει η Πρόεδρος. Το λόγο έχει τώρα η Βερόνικα Νίλσον. Πριν όμως της δώσω το λόγο, θέλω να πω ότι Business Europe ήρθε εδώ για να ενημερωθεί και για την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, μάλλον τις συλλογικέ συμβάσεις και τι έγινε στην Ελλάδα με αυτές, την παρέμβαση της Τρόικα δηλαδή εκεί. Χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ η Business Europe και πρέπει να δείτε και τις αποφάσεις που πήρε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας επίσης για το ίδιο θέμα. Η κυρία Νίλσεν, ευχαριστώ. Ναι, είπε ο συνάδελφος ότι συνήθως συμφωνεί με όσα λέει ο πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς συνήθως διαφωνούμε αν και το συγκεκριμένο δεν το άκουσα, οπότε δεν ξέρω. Πάντως να θέλω να είμαι πιο προσεκτική όσον αφορά την ανάκαμψη. Αν ακούσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαν να έχει τελειώσει η κρίση και όλα πάνε καλά. Όμως, μπορεί να πάμε σε αποπληθωρισμό. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί, ότι θα έχουμε το ιαπωνικό σενάριο και εδώ. Μπορεί να συμβεί. Και πολλοί οικονομολόγοι το λένε. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ακούω ότι έχει αρχίσει η ανάκαμψη και όλα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν κατά πόσο η τραπεζική κρίση έχει επιληθεί και η τραπεζική ένωση δεν ξέρω, δεν φαίνεται να είναι τόσο ισχυρό εργαλείο όπως είχαμε ελπίσει. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα πολλοί κίνδυνοι που αλοχεύουν. Τι χρειαζόμαστε πρώτον να σταματήσει η λιτότητα. Δυστυχώς η λιτότητα δεν έχει σταματήσει. Υπάρχει πάντα ίσως όχι όπως πριν, ίσως να έχει γίνει κάπως πιο ήπια, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει λιτότητα και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, ζήτηση στην οικονομία, κάτι που δεν έχουμε. Μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, αλλά μιλάμε για πολύ μικρά ποσά. Ποσότητες, ποσοστά. Δεν θα βοηθήσει αυτό να αλλάξει η κατάσταση, να έχουμε πλήρη απασχόληση και πάλι. Πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομία. Έπρεπε να είχα μαζί μου και τα έγγραφα των ε, συνδικάτων μας που συμφώνησαν πέρυσι τα μέλη μας με ένα σχέδιο επενδύσεων, πώς θα δώσουμε νεόθεση στις επενδύσεις, τι ε, ποσοστό του ΕΠ πρέπει να πηγαίνει σε επενδύσεις. Αυτή είναι μια λύση που προτείνουμε εμείς για την κρίση. Πρέπει επίσης να πω σε αυτό που είπε ο Τζέιμς για το διοικητικό άχθος. Βασικά δεν συμφωνούμε. Γιατί πάλι τα εργασιακά δικαιώματα πλήττονται. Είδαμε και από αυτά που είπε η Κομισιόν πέρυσι ότι με τις προτάσεις μας θέλουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, να προσφέρουμε περισσότερη ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όμως ο κοινωνικός διάλογος δεν τηρείται. Για παράδειγμα, στα κομμωτήρια δεν πήγε καν για έγκριση στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καν διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους. Έπρεπε να τα διαβάσουμε εμείς στις ε, επίσημες ανακοινώσεις. Οπότε δεν βλέπω εγώ πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά δεν σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και επανέρχομαι στη συνθήκη. Ναι, αυτή θα ήταν μια λύση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή να πάρει νομική δράση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί δεν δίνουν τη σημασία που πρέπει στη συνθήκη και στα δικαιώματα των εργαζόμενων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει η Κομισιό να γίνει και πάλι θεματοφύλακας των συνθήκων. Όσον αφορά τις συστάσεις μας τώρα θέλουμε να γίνει αναθεώρηση του μνημονίου, των μνημονίων ώστε να τηρούν τα κοινωνικά δικαιώματα και να έχουν διαφορετική οικονομική προσέγγιση. Επίσης, στο μέλλον θέλουμε ό,τι η μέτρο προτείνεται να ελεγχθεί καλά, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ευθυγραμμίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και δεν είναι αντίθετο με αυτά. Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υπάρχουν ακροάσεις με τα κοινοβούλια, κάθε φορά που προτείνονται μέτρα τύπου μνημόνια Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης θα έπρεπε να κάνει μια έκθεση προσπαθώντας να εντοπίσει όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουμε και άλλες προτάσεις. Αλλά εντάξει, έχει περάσει ο χρόνος μου. Να, αυτή είναι η έκθεσή μας. Πάρτε ένα αντίγραφο παρακαλώ για να την μελετήσετε. Ευχαριστώ. Παίρνουμε... Να ακούσουμε τώρα τις άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Πουπάκης, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικέ ε, τη Τρόικα ταυτίστηκαν με την ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων δημοσιονομική εξηγίαση και εσωτερική υποτίμηση. Υιοθετήθηκε λοιπόν ένα μοντέλο μονοδιάστατη και ακραία λιτότητα με όρου βία προσαρμογή, καταργήση λιγοριστικών συμβάσεων, νομοθετικά μείωση μισθών συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα. Και το ξέρω προσωπικά γιατί εγώ είχα υπογράψει πριν έρθω εδώ την τελευταία συλλογική σύμβαση εργασία κατώτερου μισθού. Είναι δυνατόν λοιπόν μια ερώτηση το μοντέλο αυτό να αγνοεί τι εθνικέ ιδιαιτερότητε, τι ζωτικέ κοινωνικέ ανάγκε όταν η φτώχεια εξαπλώνεται, οι κοινωνικέ δαπάνε περικόπτονται ή να αγνοούνται οι προεκτάσει των προγραμμάτων στην απασχόληση, στην πραγματική οικονομία, πραγματική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Τώρα όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει. Τρομολογήθηκαν χωρί κοινωνικό διάλογο και αναπτυξιακό περιεχόμενο. Ρωτάω, δεν είναι όλα αυτά απόκληση από τη λογική συνθήκη της Λισαβόνας, δεν είναι εκτροσυχιασμό από τους κοινωνικούς στόχους στρατηγικής 2020. Σήμερα, όταν βλέπω την ύφεση να ξεπερνά 25% συνέπεια του ομολογημένου λάθους δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών και την ανεργία να ξεπερνάει 27%, πιστεύω και θα ρωτάω, δεν πιστεύω ότι θα, θα έπρεπε να υπάρχει μια αμυγός ευρωπαϊκή λύση με αλληλεγγύη, σεβασμό αξίε δημοκρατική διαδικασία ένωση αλλά και διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρί εξαιρέσει. Και ένα τελευταίο. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποιε θα είναι οι επιπτώσει των παρεμβάσεων τη Τρόικα στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου στο εν λόγω κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα πολύ στο να κάνω μια-δυο παρατηρήσεις στα όσα είπε ο κύριος Νουαγνόγκ για τον κύριο Κάρας. Δεν είναι σωστό το να λέτε ότι έλειπε, δεν εξετίμησε την υποσυζήτηση η υπόθεση. Εμείς ως ΕΛΚ υποστηρίζουμε τις προτάσεις, υποστηρίζουμε την ψηφοφορία το Μάρτιο. Είμαστε αρκετοί νομίζω εκπρόσωποι του ΕΛΚ εδώ. Με πολύ μεγάλο σοβαρό το αντιμετωπίζουμε αυτή την ακρόαση και νομίζω ότι ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση αυτό που ακούστηκε του συνάδελφο των Σέρστον. Και προχωρώ με μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Καταρχάς θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι αποφάσεις δεν λήφθησαν πάντα μόνο ή πάντα από την Τρόικα, αλλά στηρίζονται σε αποφάσεις της, ε, του Eurogroup. Τόσο η Τρόικα λοιπόν όσο και το Eurogroup ε, εκπροσωπούνται από τα κράτη-μέλη, ε, στα κράτη-μέλη. Άρα δεν δέχομαι να αρχίζουμε μια συλλογιστική με την οποία καταλήγουμε να μετατρέψουμε την Τρόικα σε αποδιοπομπαίο τράγο, γιατί αυτό δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Εάν θυμίσουμε πού βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια κάποια κράτη ενώπιον του φάσματος της ε, χρεοκοπίας και ότι χωρίς τη βοήθεια πολλών από εμά αλλά και της Τρόικας συγκεκριμένα δεν θα ε, βρίσκονταν ίσως ε, στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα και βεβαίως πρέπει να γίνεται η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει πάντως να υπενθυμίσω ότι θα είχαν χαθεί όλα τα κοινωνικά κεκτημένα των κοινωνικών εταίρων σε περίπτωση χρεοκοπίας κάποιου κράτους. Ερωτώ λοιπόν και για το μέλλον τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι συνάπτοντας συμφωνίες με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και ποια θα ήταν τα καλύτερα μέσα για να μην υπάρξουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, ώστε ακριβώς να αποφύγουμε, ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι, ευχαριστώ, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιες κρίσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ Σαριά και Γκίγκολτ μετά. Κύριος Φαγιώ επίσης θέλει να λάβει το λόγο. Θέλω και εγώ να καταθέσω κάποιες ερωτήσεις. Κάποιος άλλος. Ζητεί το λόγο. Καλώς. Άρα, ακούμε τους, ε, θα ακούσουμε τις έξι ερωτήσεις αυτό το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης. Θα ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας και μετά αφήνω τους εισηγητές να τοποθετηθούν πριν κλείσει η συνεδρίαση. Εσαϊά, Γκίγκολτ, όπως είπαμε, για τη ζήτηση δευτερολογία και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημά μου αφορά την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες που έχουν υποφέρει περισσότερο λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες είναι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης και πληρώνουν και τους περισσότερους φόρους γιατί σπάνια μεταφέρουν ε, τα κέρδη τους σε οικονομικούς παραδείσους, φορολογικούς παραδείσους εκτός των χωρών τους. Στην Επιτροπή είχαμε μια ακρόαση που ακούσαμε ότι για παράδειγμα στην Πορτογαλία υπήρξε δραματικός αριθμός πτωχεύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, εσείς ε, πιστεύετε πως τώρα χάνουμε τη δυνατότητα για ανάκαμψη μακροπρόθεσμα διότι αυτές οι μικρομεσαίες δεν υπάρχουν πλέον ε, και ελπίνουμε πως όταν θα υπάρξει μια θετική καμπή στην οικονομία οι μικρομεσαίες σαν αυτές που θα πάρουν τη θέση τους και θα προσφέρουν θέσεις απασχόλησης. Αν όμως δεν υπάρχουν, τι θα γίνει. Ε, εσείς βλέπετε λοιπόν, θεωρείτε ότι θα πρέπει να τονιστεί η κατάσταση των μικρομεσαίων όταν συζητάμε την έξοδο από την κρίση. Εγώ Θεωρώ πως ναι, φυσικά είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, τι δικαιώματα θα έχουν εργαζόμενοι θα είναι άνεργοι, δεν θα μπορούν να προσφέρουν καμία θέση επασχόληση σε κανέναν. Νομίζω πως οι μικρομεσαίες πρέπει να έχουν κύριο ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σβέν Γκίγκολ και μετά ο Διέγκο Φέιο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το ερώτημά μου απευθύνεται στην Business Euro όσον αφορά τα θέματα παράβασης του νόμου, παραβίασης του νόμου. Αν κατάλαβα καλά, την ETUC έλεγαν ότι οι συλλογικέ διαπραγματεύσει έχουν σημαντικά περιοριστεί ε, και αυτό είναι ε, ε, σε κατά παράβαση των υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Και σέβομαι βέβαια αυτό που είπατε ότι δεν είναι μόνο η Τρόικα και, αλλά και οι χώρε αντίστοιχα πρέπει να μεταρρυθμίσουν. Εμείς όμω εδώ είμαστε για να ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν μέρη την ΕΚΤ, αλλά περισσότερο την Κομισιόν στο ρόλο τη, η οποία συνέβαλε σε αποτελέσματα τα οποία πιθανότατα είναι παράβαση της νομοθεσίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ειδική προστασίας της ανεξαρτησίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την άποψή σας από αυτού και αν λέτε ότι δεν μπορείτε να το σχολιάσετε με λεπτομέρειες εδώ, θα, πολύ θα μου άρεσε αν η Business Europe έβαζε, έδ, μας έδινε γραπτό στα σχόλιά της για αυτές τις κατηγορίες κατά ε, για την παραβίαση της νομοθεσία, γιατί αυτό αφορά την ανεξαρτησία των κοινωνικών εταίρων. Θα ήθελα λοιπόν πολύ να ακούσω την άποψή σα για το θέμα αυτό. Ο Ντίγκο Φέιο, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές για την παρουσία του σήμερα εδώ. Μας έδωσαν διαφορετικές και ενδιαφέρουσες απόψεις για τη δουλειά μας, ανεξάρτητα αν ε, συμφωνούν ή διαφωνούν. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας, ε, έχουμε την ιδέα ότι αυτή η Τρόικα προέκυψε ως επίγουσα λύση απέναντι σε πολύ ε, ε, ε, σοβαρές καταστάσεις σε ορισμένα κράτη που ήταν σε απόλυτη ανικανότητα αδυναμία να πληρώσουν τις ευθύνες τους. Ποια, θα έπρεπε να γίνει ίσως κάποια μελέτη για το ποιες θα ήταν οι κοινωνικές επιπτώσεις και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της οικονομίας εάν δεν είχε βρεθεί αυτή η λύση. Πώς θα αντέχαμε στην Ευρώπη αν δεν είχαμε σκεφτεί αυτή τη λύση. Έπειτα συγκεκριμένε ερωτήσεις για κάθε από τους δύο ομιλητές σύντομα όσον αφορά την εκπρόσωπο των συνδικάτων. Θα ήθελα να γνωρίζω τι ρόλο αποδίδει στις, ε, στις ε, συμφωνίες ε, στα κράτη όπου έχει παρέμβει η Τρόικα ε, και που θα βγουν σε λίγο από τα προγράμματα. Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις συμφωνίες ε, γιατί αυτές συνέβαλαν πολύ στην... Ε, στο καθησυχασμό της κοινωνίας μας. Έπειτα, πώς βλέπετε αυτούς τους δείκτες εμπιστοσύνης, αυτά τα μηνύματα μάλλον εμπιστοσύνης που φαίνεται να προκύπτουν για τις διάφορες οικονομίες. Εγώ είδα εδώ να γίνονται αναφορές σε αναρρύθμιτες σε μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μου, αυτό ε, δεν είναι ε, αλήθεια. Υπάρχει μια προοπτική ανάπτυξη στην οικονομία μας και θα ήθελα να ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό το ίδιο φαινόμενο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να θέσω τρεις ερωτήσεις στους προσκεκλημένους μας. Ε, η πρώτη είναι η εξή. Κάναμε έκκληση για να στηρίξουμε, τη, να τη η Τρόικα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, επειδή είναι πυρογνώμων ε, και επειδή έχει κάνει αναλύσεις για διάφορε χώρε πυρογνωμοσύνε, οι οποίες δεν ε, ήταν ε, ίσως οι καλύτερες. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, γιατί οι συμβάσεις αυτές αποτελούν μια βάση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο. Ωστόσο δεν επικαλεστήκαμε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη για να μπορέσουμε να ε, πλαισιώσουμε την εργασία της Τρόικα. Πιστεύετε πως είναι αυτό σφάλμα και αν και δυστυχώς οι πολιτικές ε, ε, ε, συζητήσεις λένε ότι θα έπρεπε αυτό, η Τρόικα να έχει πλαισιωθεί και από το διεθνέ Γραφείο εργασία. Έπειτα, εκεί όπου οι χώρε στις χώρες όπου οι μεταρρυθμίσει πάνε καλά, βλέπουμε ότι είναι χώρε όπου ο κοινωνικό διάλογο βρίσκεται στην καρδιά τη μεταρρύθμιση και όπου όλη αυτή η διαδικασία που αντιστοιχεί ακριβώ στην ευρωπαϊκή σκέψη, η ιδιοποίηση δηλαδή των μεταρρυθμίσεων από του κοινωνικού εταίρου, λειτουργεί χάρη στην ξέρω το κοινωνικό διάλογο. Πώ μπορούμε λοιπόν να έχουμε από τη μια πλευρά αυτή την αντίληψη για τη τη θέση και το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου όσον αφορά τις ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και να φανταστούμε ότι η Τρόικα μπορεί να στεφθεί με επιτυχία ε, από τη στιγμή που όσον αφορά μάλλον μια πραγματική συμβολή στην εξισορρόπηση και τον εξυγχρονισμό των χωρών. Ε, Τέλο, όταν βλέπουμε το δρόμο προ μια πραγματική ΟΝΕ, ναι, Οικονομική και Νομισματική Ένωση παντού, υπάρχουν, ακούγονται ωραία λόγια όσον αφορά τη θέση του κοινωνικού διαλόγου, του ζωντανού κοινωνικού διαλόγου και σε, και σε ευρωπαϊκό και κλίμακα. Δεν είναι όμω μια ριζική αντίθεση ανάμεσα σε αυτή την έννοια της ε, αύξησης της σημασίας και της αξιοποίησης του κοινωνικού διαλόγου και της πραγματικότητας του τι έκανε δηλαδή η Τρόικα σε κάθε ένα από τα κράτος μέλη όπου παρενέβη. Ε, αγνοώντα του βασικού κανόνε, όχι μόνο του ευρωπαϊκού, όπω διαπίστωσε το Συμβούλιο τη Ευρώπη, αλλά και τι βασικέ συμβάσει του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζει μάλλον η Business Europe, αλλά μάλλον το άκουσε σήμερα. Καλά. Ποιο από του δύο θα ήθελε να πάρει πρώτο το λόγο. Κύριε Ευχαριστώ για τις παραβιάσεις στην νομοθεσία. Εδώ ήμουν κάπως επιφυλακτικός και είναι επειδή δεν είμαι αρκετά καλά ενημερωμένος, αλλά σημείωσα τόσο είπε ο Κρυγκό που λέει ότι θα υπάρχουν, ε, λέτε, παραβιάσεις και καταγγελίες. Οπότε ε, ήμουν επιφυλακτικός ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί υποθέτεται. Οι επιχειρήσεις, οι υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι υπέρ της στήριξη του νόμου. Αυτό είναι κάτι γενικό. Αλλά φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα να έχετε μια απάντηση από την οργάνωσή μας και θα επανέλθουμε σε αυτό πολύ συγκεκριμένα αργότερα. Κάτι άλλο τώρα στο οποίο αναφερθήκατε κάποιοι από εσά, πόσο μεγάλη σημασία δηλαδή έχει ο κοινωνικός διάλογος γενικά και επιστήνεται την προσοχή μας στις εμπειρίες που έχουμε με την Τρόικα. Πολύ καλά ήταν τα σχόλια που κάνατε όσον αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες με τις οποίες ασχολούμαστε και το είπα και εγώ στην παρουσίασή μου αρχικά. Πολύ σωστό επίσης αυτό που είπατε για τη σημασία που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, χρειάζονται ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να έχουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά χρειάζεται και ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάτε για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ναι, Επί του παρόντος πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, τρόπους, βάζοντα τη φαντασία μας να δουλέψει, ώστε να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση. Και έρχομαι και σε αυτό που είπατε και εσεί γενικά για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και εδώ ναι, συμφωνώ ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά δεδομένου και του προβλήματο με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουμε βγει ακόμα από το πρόβλημα, ακόμα υπάρχει κίνδυνος. Άρα δεν μπορούμε να καθησυχαστούμε και να παρετηθούμε από το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων έτσι όπως πρέπει αυτές να γίνουν. Τι θα γινόταν αν δεν είχε παρέμβει η Τρόικα. Όταν γράφεται την έκθεση αυτή, πρέπει να έχετε ακριβώς αυτό μπροστά σας. Ότι ναι, συμφωνώ, η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη, όλοι συμφωνούμε ότι η απασχόληση δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά ακριβώς αυτό, περί αυτού πρόκειται, πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε παρέμβει η Τρόικα. Βερόνικα Βότσον. Ευχαριστώ. Έγιναν διάφορα σχόλια για το ότι είχε να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση η Τρόικα, χώρες που βρισκόντουσαν στα όρια της χρεοκοπίας κλπ. Έχω διαβάσει διάφορα μνημόνια και αναφέρονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση θέλουν οι χώρες αυτές δηλαδή να προχωρήσουν σε ελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση. Επίσης το μνημόνιο για την Κύπρο διάβασα. Εκεί υπάρχουν λεπτομέρειες για τον χρόνο εργασίας των αυτοπασχολούμενων σε νοσοκομεία για την ασφάλεια, για την υγιεινή. Γιατί πρέπει να ανακατεύεται με τις ώρες εργασίας η Τρόικα του προσωπικού στα νοσοκομεία, για παράδειγμα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Λέτε ότι η Τρόικα βοήθησε να μην χρεοκοπήσουν οι χώρες αυτές. Ναι, αλλά ίσως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι από τους οποίους θα μπορούσαν να είχαν υποφερθεί πολύ περισσότερο οι χώρες αυτές. Τώρα, ε, ρωτάτε για το κατά πόσο πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν στις συλλογικές συμβάσεις. Ναι, αλλά πια στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται αυτό, για παράδειγμα. Το Διεθνέ Γραφείο Εργασία έχει οργανώσει διάφορες συναντήσει με την Κομισιόν. Συμμετείχα και εγώ σε μία στην Αθήνα και ο Γενικό Γραμματέας τι είπε, είπε ναι, συλλογικές συμβάσεις ε, στο μέλλον θα πρέπει να είναι όχι απαραίτητα για τους μισθούς και το χρόνο εργασίας, αλλά για τη μεταρρύθμιση, νέα μέτρα, καινοτομία κτλ. Μα όχι, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τελικά η Τρόικα μας εμποδίζει να συμμετέχουμε στις συλλογικές συμβάσεις και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι διαφορετικές μεταξύ τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το τελευταίο καιρό το λέμε αυτό τόσο πολύ ότι χρειάζονται ειδική μεταχείριση γιατί αυτές δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Είναι σαν να λέμε άρα δεν χρειάζεται πια καμία ρύθμιση για αυτές. Τις αφήνουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν θα έπρεπε. Ο νομοθέτης πρέπει να αποδείξει γιατί πρέπει το θέμα των τιμών να συμπεριλαμβάνεται για παράδειγμα. Και δεν πρέπει να είναι έτσι. Οι μικρές επιχειρήσεις, όχι απαραίτητα μικρομεσαίες, αλλά οι μικρές δεν δημιουργούν και τόσε θέσει απασχόλησης. Α είμαστε πιο προσεκτικοί λοιπόν όταν μιλάμε για τι διαφορές που έχουν μεταξύ του και γιατί χρειάζονται μεγάλη προστασία. Ο ρόλο του Διεθνούς Γραφείου εργασία είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μερικέ φορέ οι συνδίκες εργασία είναι πάρα πολύ κακέ. Έχει συνεισφέρει ε, το Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και στις εκθέσει που εκπονήσατε. Τέλος, κύριε Πέρες, όσον αφορά την αντίφαση ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ δεν βλέπω την αντίφαση, γιατί δεν βλέπω καν η Κομισιόν να στηρίζει τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη. Ε, φοβάμαι ότι δυστυχώς η ίδια είναι η κατάσταση και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση αυτή που είχαμε από κοινού οι δύο επιτροπές, οικονομική και η απασχόλησης. Είναι μια δουλειά που θελήσαμε να κάνουμε για να έχουμε τον απολογισμό του έργου της Τρόικας. Ο κοινωνικός διάλογος είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχει πάντα συνένεση, γι' αυτό πρέπει να αξιολογείται από τους νομοθέτες από κοινού με τα άλλα σημεία όπως είναι η οικονομική και η κοινωνική διακυβέρνηση. Πριν ολοκληρώσουμε πάντως αυτή την ακρόαση, έχω να προτείνω οι τρεις εισηγητές να πάρουν το λόγο, δύο λεπτά ίσως ο καθένας, για να πούνε ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν μετά την ακρόαση αυτή και ποια είναι τα προσωρινά τουλάχιστον συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε πριν έχουμε βέβαια την τελική εκδοχή της έκθεσης. Εκ μέρου τη Οικονομική και Νομισματικής Επιτροπή, ο κύριος Λιαμνιόκ, παρακαλώ. Και μετά ο κύριο Ζάλμπα, εκ μέρου του κύριου Κάρας. Παρακαλώ, Λία, μέχρι το λόγο. Ευχαριστώ. σου, δεν θα συνεχίσω την αντιπαράθεση. Χαίρομαι πάντως που η ακρόαση έλαβε χώρα, εν τέλει, και που μπορούσε να εκφραστεί και η γνώμη της Επιτροπής των Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η ακρόαση, γιατί όπω βλέπουμε ότι ε, όπως βλέπουμε δεν συμφωνούν προς τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και κυρίως τις οικονομικές του συνέπειες οι προσκεκλημένοι. Σημειώνω ότι η κυρία Νίλσον μας είχε πει και σωστά ότι τα ποστά της, ε, του δανεισμού είναι σημαντικότερα, υψηλότερα από την περίοδο πριν να αρχίσει το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για τις χώρες. Άρα το πρόβλημα που προϋπήρχε δεν έχει αντιμετωπιστεί. Για τους πολλαπλασιαστές λυπούμε που ο κύριος Γότσον ε, έκρινε σκοπό να μην μου απαντήσει. Άρα καταγράφω ότι δεν υπάρχει θέση και δεν έχουν στοιχεία η ε, Business Europe. Ούτε άλλα στοιχεία μου δίνεται για την απασχόληση, γιατί μου δίνεται ένα σχετισμό μεταξύ ε, κόστος μονάδας εργασίας και κόστος απασχόλησης ε, και κόστος ανεργίας. Άλλωστε όμως ε, θα απαντήσω ότι η σχέση αυτή μπορεί να διαβαστεί και διαφορετικά. Επειδή υπάρχει ψηλή ανεργία, πουλάνε λιγότερο επιχειρήσεις και επειδή πουλάνε λιγότερο έχουν υψηλότερο κόστος απασχόλησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε στα δύο λεπτά που μας μένουν να λύσουμε τέτοια θέματα. Παραμένουν οι διαφωνίες, είναι προφανές, στους μελλοντικού μηχανισμούς αρρωγής υποστηρίξης που θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί για την Τρόικα η οποία προφανώς θα πρέπει να διαλυθεί διότι δεν έχει νομική βάση. Στη θέση της λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει νέους μηχανισμούς, θα πρέπει να επιτραπεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. Περισσότερη δημοκρατία σημαίνει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και ελπίζω ότι σε αυτό θα καταλήξει μεταξύ άλλων η έκθεσή μας σε συμπέρασμα. Ευχαριστώ κύριο Σόλμπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Καράς λυπάται που δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ σήμερα. Οπότε το μόνο που θα κάνω είναι να υπογραμμίσω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει για το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, περισσότερος κοινωνικός διάλογος δεν θα ήταν ε, θετικός για την λήψη αποφάσεων. Κάθε άλλο. Είναι αλήθεια επίσης, όπως ακούσαμε, οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες περισσότερο υπέφεραν από την κρίση αυτή. Και επιπλέον μάλιστα οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι καταδικασμένες να αποτελούν το βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάκαμψης. Είναι εκείνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου για την οικονομική ανάκαμψη. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την ενδιαφέρουσα ακρόαση. Τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ο κύριος Σέρκας, εκ μέρους Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ζητήματα ε, Πρώτα απ' κανένας δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζονται προγράμματα βοήθειας στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Εννοείται το θέμα είναι με ποιο τρόπο τα προγράμματα αυτά τίθενται σε εφαρμογή. Επίσης υπάρχει συμφωνία για το ότι οι συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές ήταν δραματικές. Σε αυτό συμφωνούμε. Εκεί που δεν ξέρω αν συμφωνούμε είναι στο τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε αυτή την ε, διάσωση από την Τρόικα ή πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Δύσκολα μπορεί κανείς βέβαια να κάνει προφητής, ο καθένας έχει τις δικές του πεπιθήσεις, πάντως γι' αυτό δεν συμφωνούμε. Η Επιτροπή πασχολησης μελετάει βέβαια τις κοινωνικές συνέπειες. Τώρα όμως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια ελπίδα για ένα διαφορετικό μέλλον από τα τελευταία πέντε χρόνια που ζήσαμε. Και για να το πετύχουμε αυτό, μια που όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια νέα εποχή, ότι δεν έχουν λυθεί ακόμα τα προβλήματα, ίσως ήρθε η στιγμή για διόρθωση και για να επανέλθουμε στα επίπεδα απασχόλησης που θέλουμε, να υπάρχει ρευστότητα, να διορθωθούν οι κοινωνικές αδικίες, αυτά να αλλάξουν. Και γι' αυτό για την Επιτροπή μας τουλάχιστον αυτό που ισχύει είναι ότι ο στόχος μας είναι το μέλλον. Είναι μια γενιά που στην Νότια Ευρώπη έχει καταστραφεί. Και η καταστροφή είναι διαρθρωτική, δεν είναι συγκυριακή πια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στην ακρόαση όπως είπαμε και στην αρχή, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε όλη αυτή τη διαδικασία εξέτασης των αποτελεσμάτων από τις δράσεις της Τρόικας. Ο καθένας τώρα θα καταλήξει στα συμπεράσματά του μετά από την ακρόαση αυτή για να συνεχίσει τη δουλειά του είτε πρόκειται για την Οικονομική Επιτροπή είτε για την Επιτροπή Απασχόλησης. Και θα τα πούμε και στην Ολομέλεια βέβαια γι' αυτά. Ωραία, έληξε η κοινή αυτή ακρόαση. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας αφήνουμε τώρα την Οικονομική Επιτροπή να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ.